Καλημέρα, ξεκινάει η σύνοδος. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τον κανόνα ε, της ε, μοναδικής χειραποσκευής που επιβάλλουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Ο κύριος Σίμψον, που είναι ο συγγραφέας, έχει πέντε λεφτά για να μας παρουσιάσει την ερώτηση. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε ήδη, γιατί δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Επιτροπής. Αξίζει τον κόπο.